να στέλνουμε μηνύματα σαφέστατα όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Πεντεχούχτ. Ε, ο συνάδελφός ο κύριος Μπρόκ έχει τώρα το λόγο ως πρώτος ομιλητής από τα πολιτικά κόμματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι.